Περνάμε τώρα στις ε, επεξηγήσει ψήφου. Και ο συνήθως ε, θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους να εγκαταλείψουν την αίθουσα ησύχως. Und für diejenigen, die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 Περνάμε τώρα στις ε, επεξηγήσεις ε, ψήφου. Είχαμε λάβει πολλά αιτήματα αν δεν καταφέρουν όλοι να μιλήσουν θα ήθελα να σας πω πως θα πρέπει να διακόψουμε για να μπορέσει να συνεχιστεί η συνεδρίαση το απόγευμα. Λοιπόν, περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ε, ψήφου. Όχι, όχι, πρώτα ε, θα ακούσουμε τον συνάδελφο επί της διαδικασίας. Κύριε Πρέιδρε, εδώ τι είναι σύλλογο συζήτηση φοιτητών ή κοινοβούλιο. Μιλάμε για σοβαρά ζητήματα. Είχαμε όλοι συμφωνήσει στο ΕΛΚ και τους φιλελευθέρους, ε, ενώ και το κείμενο τελικώς άλλαξε τελευταία στιγμή. Ακόμη δεν καταλαβαίνουμε σε ποιο κείμενο ακριβώ, επί ποιο κειμένου ψηφίζουμε. Αλλά μιλάμε για μια ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη και βλέπουμε δύο πολιτικέ ομάδε ε, το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες να εκβιάζουν ε, την κατάσταση και να αποφασίζουν αν θα αναβληθεί το κείμενο ή όχι η ψήφιση μάλλον για ένα δεκαπενθήμερο. Δεν υπάρχουν επαρκείς εξηγήσει και δεν ξέρουμε τελικά τι ψηφίζουμε. Δεν είναι αυτό δημοκρατία κύριε Πρόεδρε. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ε, θα έπρεπε επιτέλους ήρθε η στιγμή να το αποφασίσουμε και σε αυτό το σώμα. Συνάδελφε, σας διαβεβαιώ, δεν είμαστε φοιτητική συνέλευση. Είμαστε δημοκρατία, γι' αυτό ψηφίσαμε. Η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της αναβολής. Αυτό ήταν η μία περίπτωση που αναφέρατε. Στη δεύτερη, η ομάδα σας είχε την ευκαιρία να μιλήσει. Ρώτησαν κάποιος ήθελε ε, να πει κάτι για την τροπολογία της κυρίας Λούνατσεκ. Δεν σηκώθηκε κανείς. αν υπήρχαν αντιρρήσεις. Κανείς δεν έβγαλε κύχ. Ούτε κι εσείς μπορούσατε να το πείτε. Άρα ψηφίσαμε όπως ήταν το αίτημα σύμφωνα με, τους, με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ αγαπητέ. Και... Πρόεδρε, δεν ήταν όμως σαφές τι θα ψηφίζαμε ή τι δεν θα ψηφίζαμε. Δεν καταλάβαμε τελικά ποιο ήταν το κείμενο. Συνάδελφε, υπάρχει για κάθε θέμα εδώ πέρα ένας αρμόδιος από κάποια κοινοβουλευτική ομάδα. Και συνήθως σηκώνει το χεράκι πάνω ή κάτω αν δεν είστε σίγουρος πως πρέπει να ε, ψηφίσετε. Αν ε, δεν συνέβη αυτό δεν ε, φταίω εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με τις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση πρόοδου 2015 Σερβία σε Thank you very much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 Ευχαριστώ. Οι διαπραγματεύσεις καλές είναι με τη Σερβία, όμως ε, ελπίζουμε ούτως ή άλλως να συνεχίσουν και οι διαπραγματεύσεις με άλλες βαλκανικές χώρες. Ποιο είναι το πρόβλημα, είναι ότι αμφιταλαντευόμαστε, δηλαδή ε, θεωρούμε ότι άλλα μέτρα μπορεί να ισχύουν για την, ε, και σταθμό μπορεί να ισχύουν για τη Σερβία και άλλα για άλλες χώρες. Αφήνουμε τη Ρωσία να επικρατεί στη Σερβία, στην σερβική αγορά, να ασκεί πιέσει μέσω της Σερβία. Κάνουμε κοινέ στρατιωτικές ασκήσεις ε, με τη Ρωσία και αυτό που θέλουν να ε, διαλύσουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στην έκθεση να ξεκαθαρίζουμε ότι θα πρέπει η Σερβία να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι και η θέση της ε, χώρα. Θα πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Σερβία να αποκοπεί, να απογαλακτιστεί από την Ρωσία. Πρέπει επί να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προτού προχωρήσει. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να, ε, εμείς να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και να βοηθήσουμε τη Σερβία να το πετύχει αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Σελίμωβιτς. Χάναν. Ευχαριστώ κύριε του Πρόεδρε. Σίγουρα ήταν πολλά τα βάσανα αυτή της μεγάλης χώρας ε, στο παρελθόν ε, και ε, από το 32 όταν άρχισε με τους λιμούς ο Σταλίν και το 44 όταν έφυγαν τα τελευταία στρατεύματα ήταν η πλέον επικίνδυνη περιοχή στον κόσμο που μπορεί κάποιος, μπορούσε κάποιος να βρεθεί και ακόμη και με αυτά τα μέτρα και στεθμά οι ταταρί της Κρυμαίας έχουν υποφέρει περισσότερο από άλλους την περασμένη φορά που ήμουν στην Ουκρανία συναντήθηκα με ανθρώπους που μας περιέγραψαν αυτά που λέμε στην έκθεση περιορισμό της ελευθερίας σκέψη ανεξιθρησκείας, βασανιστήρια απαγωγές ε, και ούτω καθεξής. Ε, πώς μπορεί ε, το Κοινοβούλιο να επεμβαίνει σε αυτή την απομακρυσμένη χώρα. Αυτό είναι άλλο θέμα, άλλο Ευαγγελιο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τελικά σε ποιο στρατόπεδο είμαστε, γιατί κάποιοι εδώ μέσα ουσιαστικά βρίσκουν δικαιολογία ε, για τον ε, Πούτιν. Να μας πούνε σε ποιο στρατόπεδο είναι. Κύριε Χάναν, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά αφορούσαν τη Σερβία. Ε, έχετε βέβαια ζητήσει και τον λόγο για ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πώς πεισή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα αυτή την έκθεση για την Σερβία. Είναι προ συμφέρον της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να προσχωρήσει αυτή η χώρα. Όμως ε, θα πρέπει να πληρούνται πολιτικές ε, προϋποθέσεις για τη δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα. Φυσικά υπάρχει πρόοδος, όμως σίγουρα διαπιστώνονται ακόμη σοβαρές ελλείψεις και θα πρέπει να τις υποδείξουμε και να ξέρουμε πού ακριβώς ε, θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. Στον τομέα της δικαιοσύνης πόρο απέχουν από το κράτος δικαίου, από το ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα. Θα πρέπει να θεσπιστεί η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος τι θα γίνει επίση με την ανεξαρτησία από τη Ρωσία. Δεν μπορούν να έχουν τόσο στενού δεσμού, με τη Ρωσία αν θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επανειλημμένα να το τονίζουμε Σας ευχαριστούμε. Ε, κύριε Πολμπίση, Μαμίκινη τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν απλά στι σχέσει Σερβία Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε να δούμε ε, τι γίνεται με τον αμφίλιο πόλεμο, τι ιστορικέ μνήμε και του βομβαρδισμού του ΝΑΤΟ στη χώρα αυτή. Η εξομάλυση των σχέσεων με τι γειτονικέ χώρε βεβαίω και οι δύσκολε σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία δεν διευκόλυναν την όλη κατάσταση. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για τη ζωή τη Σερβία σήμερα και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τη βελτίωση τη κατάσταση για τι ερχόμενε δεκαετίε. Η Σερβία παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει ενεργά να εφαρμόζει μεταρρυθμίσει προκειμένου να συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό. Ε, το ίδιο και στον, ε, στο επίπεδο τη νομοθεσία. Η Σερβία αυτή τη στιγμή έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και στην κρίση των προσφύγων, λαμβάνοντα υπόψη τη σημερινά προβλήματα και του διαθέσιμου πόρου τη και προτού προσχωρήσει βεβαίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, σαφείς επιλογές. Πάντως δεν μπορώ να φανταστώ τα Δυτικά Βαλκάνια χωρίς την Σερβία. Ευχαριστούμε κύριε Μαμίκιν. Ο κύριος Γιάρ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα την έκθεση αυτή γιατί θεωρώ πως είναι ισορροπημένη. Είναι καλό το ότι συζητάμε ο με τον άλλον πρέπει να ρίξουμε φως στην υπόθεση, χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία, μιλάμε για θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, θέλουμε να αυξήσουμε και το επίπεδο ζωής των ανθρώπων, υπάρχουν και κάποιες σκίες, αλλά μπορούμε να το πούμε και ως εξή νομίζω αυτά θα μας οδηγήσουν στο να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με τους Σέρβους και δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε αμέσως με τη διαδικασία της ένταξης. Ξεκινάμε με συνομιλίες, με τις κοινέ αξίες, με την κοινή ευθύνη για αυτή την Ευρώπη. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ πως δεν είναι η τελευταία έκθεση πρόοδο, αλλά χαίρομαι για την περαιτέρω συνεργασία με τη Σερβία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία αυτή. Σας ευχαριστώ η κυρία Γεσοβιέτσκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπωσδήποτε το 2015 ήταν ένα έτος σημαντικό για τις σχέσεις με τη Σερβία. Μετά από τρία χρόνια συνομιλιών ε, μετά από τρία χρόνια ξεκίνησαν οι συνομιλίες με συγχωρείτε οι ενταξιακές ε, αλλά Βεβαίω, υπήρχε και μια επικοδομητική στάση της Σερβίας απέναντι στις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα το Κωσφοπέδιο και την στάση της κυβέρνησης κατά τη μεταναστευτική κρίση. Στήριξα την έκθεση γιατί οι αποφάσεις του Βελιγραδίου μας προστάτευσαν από μια ανθρωπιστική καταστροφή. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως η χώρα αυτή αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τα εσωτερικά της συστήματα οι διαπραγματεύσεις μόλις ξεκίνησαν δεν θα είναι εύκολες αλλά υπάρχει και άλλο ένα θέμα που δεν μοιάζει να το έχουμε συζητήσει αρκετά είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες που έρχονται στην Σερβία και την Νορβηγία και είναι Σέρβοι πολίτες φαίνεται πως η κατάσταση η οικονομική είναι δύσκολη και πρέπει να βελτιωθεί σας ευχαριστώ κυρία Κεσοβιέτσκα. Τελείωσε λοιπόν η έκθεση προόδου. Ακολουθούν τώρα τα ψηφίσματα για το πεδίο. Ο κύριος Χάναν λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κάτι τράβηξε την προσοχή μου, διότι ακόμη και από αυτά που περιμένω πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση μου κάνει εντύπωση. Αποκάλυψε από ένα, ε, για ένα βασικό ε, σκάνδαλο στο Κωσυφοπαίδιο, όπου εμπλέκεται και η ίδια η αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς. Είναι δημικό φαινόμενο η διαφθορά στο Κωσυφοπαίδιο. Γιατί, για ποιο λόγο, για τον ίδιο λόγο που είναι και ενδημικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραβάμε τους κακούς. Ε, ο ε, Έλμαρ Μπρόκ παραδείγματο χαρή. Δεν θεωρώ ότι είναι κακός άνθρωπος παρότι διακόπτει όλη την ώρα μέσα στη συζήτηση. Όχι, μέχρι αποδείξεως το αντιθέτω δεν θα το ισχυριστώ όμως. Δεν ε, υπάρχει λογοδοσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εάν αυτοί που κατέχουν την εξουσία δεν χρειάζεται να λογοδοτούν στους ψηφοφόρους, τι θα κάνουν, θα βολεύονται και ε, υπάρχει ο φόβος για το διχασμό. Δεν θέλουν να αναγνωριστεί το ελεύθερο κράτος και γι' αυτό αυτοεξυπηρετείται αυτό το διεφθαρμένο κράτος και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ίδια συμβαίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άτομα προσωπικότητες όπως ο Έλμα Μπροκ εκλέγονται ακριβώς αυτού του συστήματος. Ευχαριστώ. Πώς Eh, Ευχαριστώ. Είμαι από αυτούς τους πολιτικούς που πιστεύουν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο με το Κωσυφοπαίδιο, να προσφέρουμε σε αυτή τη χώρα μακροπρόθεσμη προοπτική για την προσχώρηση στην Ένωση. Παρότι το Κωσυφοπαίδιο ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί από πάνω από πέντε ευρωπαϊκέ χώρε. είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογο εάν θέλουμε στο μέλλον τελικά να εκδημοκρατιστεί η χώρα, να γίνεται σεβαστό το κράτο δικαίου και να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι μακρύ ο δρόμο για αυτή τη χώρα και τα 15-20 προσεχή χρόνια δεν πρόκειται να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κοσφοπέδιο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ε, επίσης, να, ε, ε, η και η διαφθορά, η μη καταπολέμηση τη οργανωμένη εγκληματικότητα, η παραβίαση των αρχών του κράτου δικαίου. Αυτά θα πρέπει να μα απασχολούν περισσότερο από την οικονομική ανάπτυξη. Και γι' αυτό εγώ υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα. Σα ευχαριστούμε, συναδελφέ Πολ Πρισίλ. Ο κύριο Μάμικινε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ξέρουμε ότι μονομερός αυτό ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο το κοσυφοπαίδιο και ε, πέντε κράτη-μέλη δεν το έχουν αναγνωρίσει το, το κράτος αυτό. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο πως ε, γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να περιμένουμε πλήρη εφαρμογή νομικών πράξεων ε, όσο επίσης δεν έχουν ρυθμιστεί και οι σχέσεις με γειτονικές χώρες, όπως με τη Σερβία παραδείγματος χάρη. Αυτό αναφέρεται μέσα στην έκθεση. Μην ξεχνάμε την υψηλότητα το ποσοστό ανεργίας προσπαθεί να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα. Σίγουρα έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το δρόμο που οδηγεί το κοσυφοπαίδιο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ακόμη να κάνει πάρα πολλά για να γίνει και de facto ανεξάρτητη η ε, χώρα. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Μαμικίνσε, ο Σάρφουρ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ θετικό και στη ημερήσια διάταξη το ότι μιλήσαμε πρώτα για τη Σερβία και μετά στο... για το κοσυφοπαίδιο. Βλέπουμε λοιπόν το διαμεσολαβητικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι αυτό της Ευρώπης και μας δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα δύο κράτη και θεωρώ πως πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτό τον επικοδομητικό μας ρόλο και να χαιρετήσουμε την πρόοδο στο κοσφοπέδιο και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις με τη Σερβία. Οπότε πρέπει να μιλάμε με τις δύο χώρες και το είπαν οι συνάδελφοι. Ιδιαίτερα ανησυχώ για το κοσφοπέδιο, για το ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποια κρατική διοίκηση που να λειτουργεί και πρέπει κάποτε να τελειώσει η διαφθορά. Αλλά παρόλα αυτά να μιλήσουμε με τις δύο χώρες και να συνεργαστούμε μαζί τους. Σας ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Γεια σας Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως η κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο πέρυσι επισκοπείται στην έκθεση. Θα πρέπει όμω να επικεντρωθούμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοσμοπεδίου, ώστε όλες οι εθνικές μειονότητες να γίνονται σεβαστές. Υπήρξαν βελτιώσεις λοιπόν σε κάποιους τομεί, όμως η χώρα αυτή έχει και κάποιες σοβαρές παθολογίε που θα δυσχεράνουν και την εξέλιξή της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εργασίες της Εθνοσυνέλευσης καθυστερούν. Η επαναφορά του κοσφοπεδίου στα δικά μας πρότυπα και με την αποστολή που οργανώθηκε για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτό προχωρά, διαπίστωσε μεγάλα επίπεδα διαφθοράς. Οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες ε, βλέπουν ότι το κοσφοπέδιο επί σειρά ετών παραμένει πηγή διαφόρων μορφών παράνομου εμπορίου δεν μπορεί λοιπόν παρόλα αυτά να θεθεί μόνο στην τύχη του το κοσυφοπαίδιο. Θα πρέπει να στηριχθεί το ψήφισμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει όλα τα μέσα για να αποτιμήσει σωστά τη χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να επιτρέψει σε ένα ακόμη αποτυχημένο κράτο να στέκεται στα σύνορά τη. Ευχαριστούμε. Κυρία Γεσλοβιέσκα. Ευχαριστώ. Σα παρακαλέσω να μην γράφετε περισσότερα στα κείμενά σα από όσα μπορούν να εκπονηθούν σε ένα λεπτό γιατί δεν μπορούν να σας ε, ακολουθήσουν οι διερμηνείς και σας καταλαβαίνουν μόνο οι συμπατριώτες σας και αμφιβάλλω και για αυτούς. Σελίμοβιτς. Είναι ευπρόσδεκτη η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση του Κωσυφοπέδου και ελπίζω να, ε, και όλες οι βαλκανικές χώρες σύντομα να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ε, θα πρέπει να εξομαλυνθούν και οι συζητήσεις με την μειοψηφία, τη σερβική μειοψηφία στο Κωσυφοπέδιο. Αυτό αποτελεί εκ των ε, όνου κάνεφε προϋπόθεση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε το θέμα σε συνδυασμό με τη Σερβία. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει ο διάλογος με τη σερβική μειοψηφία να είναι απαραίτητο απαραίτητη προϋπόθεση. Η αιρετή κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου έχει κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεράσει τα προβλήματα με σευρική μειοψηφία. Θα πρέπει λοιπόν να μην χρησιμοποιείται ε, για εγχώρια ζητήματα από τη Σερβία αυτή η κατάσταση στο Κωσυφοπεδίο και όλοι θα πρέπει να υπομιστούν τη δική του ευθύνη. Εγώ υπερασπίζομαι το ψήφισμα διότι εκεί τονίζεται ότι υπάρχει βούληση από πλευρά ε, του Κωσυφοπεδίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθηθεί η διαδικασία προσχώρησης. Ευχαριστούμε κύριε Σελίμοβιτς. Ε, Πόλτσακ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι πεπισμένος ότι το κοσυφοπαίδιο ε, πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο μέλλον. Γι' αυτό στήριξα αυτό το ψήφισμα. Όμως πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το, κοινο, το έχει κάνει τεράστιες ε, πρόοδους στον τομέα της μεταρρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, του δικαστικού συστήματος, όμως στον επίπεδο της απασχόλησης, του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς υπάρχουν ακόμη προβλήματα. συμμορίες πολλές φορές λιμένονται το, την επικράτεια της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα αυτή. Είναι τόσο κοντά στη σύγκληση με τι δικέ μα αρχέ και αξίε. Δεν θα πρέπει να τι επιτρέψουμε, να την εγκαταλείψουμε στην απομονωσή τη. Θα πρέπει να τη στηρίξουμε κατά τρόπο ώστε να ε, βοηθήσει ακόμη και στην επίλυση του προσφυγικού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πόλτσακ. Τελειώσαμε με το ψήφισμα ε, για το κοσίφο πέδιο. Περνάμε τώρα σε επεξηγήσεις ψήφου για την Λιβύη. Ο κύριος Άναν δεν είναι εδώ. Άρα ξεκινάει ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθε, κατά τη διάρκεια τη συζήτηση για τη Λιβύη, μίλησα για κάποια μεμονωμένα, μιλήσαμε για κάποια μονομένα φαινόμενα στη χώρα αυτή, την απαγωγή Ευρωπαίων πολιτών στην επικράτεια. Όμω ένα Τσέχο πολίτη λείπει εδώ και ένα χρόνο και δύο μήνε. Αγνοείται η τύχη του. Δεν είχα την, ε, το χρόνο να μιλήσω για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση χθε, γι' αυτό ζήτησα το λόγο για σήμερα. Στήριξα παρόλα αυτά το ψήφισμα αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό σε μια ε, κατάσταση όπου πολιτική συμφωνία έχει προταθεί για τι συγκρόμενε πλευρέ στη Λιβύη ήδη από πέρσι και δυστυχώς απορρίφθηκε από το κοινοβούλιο του Μπρουκ, τουλάχιστον ε, το ίδιο και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να υψώσει τη φωνή της στο διεθνές προσκήνιο και να καλέσει όλες τις πλευρές να σεβαστούν την κυβέρνηση αυτή, να προσπαθήσουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ώστε η εύθραυστη αυτή ε, εκεχηρία που έχει επιτευχθεί να διατηρηθεί προκειμένου να αποφύγουμε περαιτέρω επιδείνωση. Γι' αυτό καλωσορίζω το ψήφισμα αυτό και ελπίζω όλε τι πλευρέ να αναλάβουν δράση τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριε Πόσπιση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άλλο ένας χρόνος που εμφύλιος πόλεμος μένεται στην Λιβύη. Ε, εκατοντάδες χιλιάδες ε, αναγκάζονται να διαθήκουν ως πρόσφυγες. Και δεν είναι σαφές εάν πρόκειται να επιγραφεί συμφωνία ή να γίνει σεβαστή η συμφωνία της 17η Δεκεμβρίου μεταξύ ε, του ΟΗΕ και Τη Εθνοσυνέλευσης, της προσωρινής Εθνοσυνέλευσης του ε, η Λιβύη είναι μια από τι πλουσιότερε χώρε στην Αφρική και ευρύτερα στην περιοχή τη Μέσης Ανατολής. Δεν θα πρέπει βεβαίω να ξεχνάμε τα προβλήματα του καθεστώτος Καντάφη. Αυτά παραμένουν ε, και το βιωτικό επίπεδο τη χώρα παρόλα αυτά ήταν πολύ υψηλό. Αλλά ε, είχε να κάνει με τι τιμέ των καυσίμων. Αυτό το, επίπεδο, το βιωτικό επίπεδο μπορεί και πάλι να γίνει πραγματικότητα για τη Λιβύη εφόσον την βοηθήσουμε, την στηρίξουμε ε, στην, στην, ε, πάνω από την οικογένεια των δημοκρατικών χωρών. Ευχαριστούμε κύριε Μαμικίνης. Κύριε Ζιαρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα γερμανικά λέμε ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένο με καλές προθέσεις. Καλές προθέσεις είχαμε στη Λιβύη, ε, να σταματήσουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά η κατάσταση μας δείχνει ξεκάθαρα ποια λάθη ε, μπορούν να γίνουν μετά την πτώση ενός δικτατορικού καθεστώτος. Κάναμε πολλά λάθη, οπότε εμείς πρέπει τώρα που βοηθήσαμε να πέσει ο δικτάτορας ε, να βοηθήσουμε τώρα και στην ανοικοδόμηση και θα πρέπει να έχουμε και σωστούς εταίρους. Και το απίστευτο που έχουμε στην Λιβύη είναι πρώτον ότι δεν υπάρχει κράτος ε, και δεύτερον το είπε ο συνάλφος έχει πέσει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων οπότε δεν είναι καλό παράδειγμα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Τελείωσε και η Λιβύη. Περνάμε στην νησιωτικότητα. Ο κύριος Χάναν δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ. Στον κόσμο σήμερα υπάρχουν ε, πολλά, πολλές ε, νήσοι, μεγάλες, μικρές, υπηρετικές, ε, ηφαιστογενείς. Πολλές φορές αυτές που είναι μακριά από τις διάφορες υπήρους, την ξηρά έχουν δύσκολες συνθήκες να αντιμετωπίσουν, αντίξωες και κάποιες φορές δύσκολες συγκοινωνίες για την επικοινωνία ακόμη και με τη δική τους χώρα. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σαφή στην νησιωτική της πολιτική και ως προς τα προγράμματα χρηματοδότησης και την διασύνδεση των νήσων και ούτω καθεξής. Επίσης αφήνεια χρειάζεται σε ό,τι αφορά την στρατηγική ανάπτυξή τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ε, ίσως λίγο υπερβολικό βέβαια, είναι αυτό της οικολογικής καταστροφής στην ίσο Νάουρο όπου ε, το δυναμικό της νήσου δεν ε, στηρίχθηκε αποτελεσματικά, δεν αξιοποιήθηκε αποτελεσματικά. Στηρίζω το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Ευχαριστούμε κύριε Μάκη Ο κύριος, η κυρία Στήλερ. Ευχαριστώ. Οι νησιωτικές κοινότητε στην Ευρώπη παίζουν ζωτικό ρόλο και πρέπει να τι αναγνωρίσουμε. Για τις αεφόρε πηγέ ενέργειας έχουν τεράστιες δυνατότητες. Πρέπει να βοηθήσουμε τα νησιά μας να τις εκμεταλλευτούν και τα σκοτσέζικα νησιά με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον Ατλαντικό έχουν πολύ καλές ευκαιρίες. Για την εκπαίδευση, ειδικά η πρόσβαση στην ε, περαιτέρω εκπαίδευση, έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και έχουμε ένα νέο πανεπιστήμιο στην Σκοτία, το Highlands and Islands, το οποίο προσελκύει παγκόσμιο ενδιαφέρον και έρχομαι τώρα στην ψηφιακή πρόσβαση. Πρέπει να διασφαλίσουμε οι νησιωτικές κοινότητες να έχουν πρόσβαση σε γρήγορη ευρυζωνικότητα και είμαι υπερήφανη που εκπροσωπώ τις ε, νησιωτικές κοινότητες της Σκοτίας. Σας ευχαριστώ Χάρκιν. Με τα χαρά στήριξα την έκκληση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στι είσοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρξουν διευθετήσει για να αντιμετωπίσουμε την, τον αποπληθισμό και να υπάρξουν σωστέ αεροπορικέ συγκοινωνίε. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να θίξω το θέμα τη αεροπορική πρόσβαση σε τρία νησιά τη δυτική ακτή τη Ισλανδία. Του Ινσμόρ, του Ινσμάν και ενό ακόμα. Θα πρέπει ε, να ε, διατηρηθούν οι τρέχουσε διευθετήσει, διότι υπάρχει αεροσκάφο που εξυπηρετεί την επικοινωνία του με την ενδοχώρα, όμως αυτή τη στιγμή προβλέπεται ανταλλαγή τη πρόσβαση με αεροσκάφο σε σύνδεση με ελικόπτερο. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να δούμε κατά πόσον ο κανονισμό, όπου η υποχρέωση παροχή δημοσίων υπηρεσιών επιβάλλει τον όρο ΕΚΑΙ, δηλαδή αερομεταφορέας, με μια ειδική άδεια να ε, καταλήξω στο ότι η χρήση ελικοπτέρου ή αεροσκάφους είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι εθνικές αρχές. Όμως θα πρέπει να συμμορφωθούν με την κοινοτική οδηγία. Οι ε, κάτοικοι των τριών αυτών νήσων αξίζουν την παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ισχυρικότητα. Περνάμε τώρα στον ρόλο των ΟΤΑ στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Κύριος Χάναν απουσιάζει. Μάμικινς και πάλι. Ο προϋπολογισμός για το 2014-2020 είναι 454 δις ε, επενδύσεις ε, στις τηλεπικοινωνίες, ε, στα στην ενεργειακή αγορά και καταβάλλονται ποσά κυρίως ε, στην Ήπεθρο αλλά και οι αστικές ε, περιοχές ε, έχουν όλο ένα και σημαντικότερο ρόλο σε όλους τους τομείς όπου υπάρχουν πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και πέρα από το σοβαρότατο πρόβλημα της συμμετήκηση των Λιθουανών προς ε, δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η αλλά και μεγάλες αστικές περιοχές, ανακαίνιση σπιτιών, υποδομές, τηλεπικοινωνίες, ενεργειακή τροφοδοσία. Ε, χάρη στα κονδύλια του ΕΚΤΕ είμαι υπερψήφισα αυτή την πρόταση και ελπίζω να ε, συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το τόσο σημαντικό ρόλο στο τομέα αυτό. Η κυρία Στάλερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, οι περιφερειακές αρχές έχουν ζωτικό ρόλο για την ανάπτυξη των περιοχών και πιστεύουμε ότι αυτό συνιστά πλανέκτημα για τις χώρες και πρέπει να το προστατεύσουμε και γι' αυτό αποθαρρύνομαι από αυτά που συμβαίνουν στη Σκοτία βάσει της τοπικής κυβέρνησης περικόπτω τα κονδύλια για τους ΟΤΑ ε, και βλέπουμε ότι είναι 500 εκατομμύρια λίρες αυτή η περικοπή προωθήνει η τοπική κυβέρνηση και είδαμε ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να υποστηρίξει τι φιλελεύθερε προτάσει σε σχέση με την προστασία των βασικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένε περιοχέ που υποφέρουν με τι πολιτικέ λιτότητε. Προτού γίνει αυτή η περικοπή, προσπαθούμε να φροντίσουμε 600 παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν, να κάνουν και να γράψουν γιατί δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ε, έχουμε, απογοητεύουμε τα παιδιά της σκοτία. Ε, δεν μπορούμε να υπονομεύουμε το ρόλο των ΟΤΑ. Ευχαριστούμε, κυρία Στάιλερ. Ε, Κόλτσακ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι μέλος ενός κινήματος ε, στη χώρα μου που δραστηριοποιείται στους ε, ΟΤΑ. Γι' αυτό στήριξα αυτή την έκθεση. Ο ρόλος ε, των ΟΤΑ είναι πολύ σημαντικός με την επικουρικότητα. Συμμετείχαν και συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, και έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία όλες αυτές οι πολιτικές. Η κοινοτική ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια μεθοδος δοκιμασμένη, δουλεύει, λειτουργεί. Η ΜΚΟ, οι Δήμοι, οι επιχειρήσεις εμπλέκονται, οι κοινότητες. Ε, κάποιες χώρες απομακρύνονται από αυτή τη μέθοδο. Εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να κάνει μια ανάλυση για το πώς ε, μας βοηθάει αυτό. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα λοιπόν την ε, τα θέματα που αφορούν ε, πλέον τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξεκινάμε με την εξόντωση θρησκευτικών μειονοτήτων από το ΙΣΙΣ, Σκρίπεκ. Ευχαριστώ, χαίρομαι που κάναμε αυτό το σημαντικό βήμα σήμερα και αναφερθήκαμε στην σφαγή χριστιανών και λοιπόν και την ονομάσαμε γενοκτονία. Σήμερα λοιπόν τους δώσαμε ένα μήνυμα ελπίδας. Είναι ένα ιστορικό βήμα, αναγνωρίζουμε τα εγκλήματα του Ισλαμικού κράτους, αλλά τα είπαμε και με το όνομά τους, γενοκτονία. Βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει και τις συνέπειες. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας ε, στην περιοχή του Ράτζοβα όπου χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να ανοίξουν αμέσως ε, τα τουρκικά σύνορα στο Κουρδιστάν. Δύο εκατομμύρια άνθρωποι σχεδόν εξυπηρετούνται από μια συνοριακή διάβαση. Δεν μπορούμε να λύσουμε ολόκληρη την Συριακή κρίση, αλλά μπορούμε να σώσουμε δύο εκατομμύρια ανθρώπους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Χελβενή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας πω ότι έχω βαρεθεί πραγματικά να μαθαίνω ε, τα νέα από το Ισλαμικό κράτος. Έχω μεταβεί επανειλημμένα εκεί στην περιοχή και σε ό,τι αφορά τα κατεπήγοντα είναι πραγματικά κατεπήγουσα η κατάσταση και οι δικές μας διαδικασίες είναι σε ρυθμό σαλιγκαριού. Είναι έσχος αυτό το πράγμα. Τώρα ε, έχουμε επιτέλους την ευκαιρία να αντιδράσουμε και να κάνουμε κάτι χρήσιμο για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Περί αυτού πρόκειται. Μέχρι τώρα η Ευρώπη δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ούτε στις ευθύνες της απέναντι στις θρησκευτικές μειονότητες και δι' τους χριστιανούς. Μετά από χρόνια καθυστερήσεων το έχουμε καταλάβει οι θρησκευτικέ μειονότητε έχουν το βλέμμα του στραμμένο στην Ευρώπη και ελπίζουν. Ε, ε, δεν θα πρέπει να του αρνηθούμε τη βοήθειά μα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο επόμενο έδαφος Χάν αναποσιάζει, ο κύριο Πόσπισης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν υπέρ αυτού του κειμένου. Οι λόγοι έχουν εξηγηθεί από τους το Ισλαμικό κράτος δεν είναι κράτος καθόλου. Είναι μια ομάδα τρομοκρατών και είναι επομένως ε, απαραίτητο να μπορέσουμε να περιγράψουμε την δράση τους. Τη δράση τους η οποία ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια που υπάρχουν ε, ε, δηλαδή εγκλήματα της ανθρωπότητας, γενοκτονία, όλα αυτά που δημιουργήθηκαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε θα πρέπει να δούμε το πώ. θα προσαγάγουμε ενώπιν τη δικαιοσύνη του ε, επικεφαλεί του Ισλαμικού Κράτου. Τώρα και κάτι άλλο θέλω να σα πω. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να καταδικάσουμε όλε αυτέ τι πράξει ε, ε, καταστροφής του πολιτισμού και επίση θα πρέπει να καταδικάσουμε όλου ε, οι οποίοι έχουν οικονομικά συμφέροντα και υποστηρίζουν το Ισλαμικό κράτο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για ε, τα κράτη-μέλη. Να προσέξουμε να μην ζητούμε τα, τα προϊόντα αυτά γιατί αλλιώς δεν θα ωφελούνται. Ευχαριστώ. Κύριε Πόσπισε, τελευταίος ο κύριος Μαμίκινς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ανεξαρτήτως του ΕΑΟΑΙΣΙΣ ακολουθεί τους Ισλαμικούς κανόνες ή τους διαστρεβλώνει πλήρως, ε, γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι φυσιολογικοί. Κανένας από αυτούς. Αυτά που βλέπουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή δεν έχουν καμία σχέση με την ανθρωπότητα ούτε με την ανθρωπιά. Το ΝΤΑΕΣ, το Ισλαμικό κράτος, καταπιέζει και τους μουσουλμάνους. και τους, ε, τις μειονότητες χριστιανούς, γεζιτοί και άλλους ε, οι οποίοι είτε θα προσυλλητιστούν είτε θα πεθάνουν. Δεν τους αφήνουν άλλη επιλογή. Όταν δεν υπήρχε το Ισλαμικό κράτος, ε, είχαν προβλήματα, αλλά τώρα ε, κινδυνεύουν να τους εξοροθρεύσουν. Γι' αυτό είναι και πρόσφυγες περισσότεροι. Θα πρέπει να οργανώσουμε ε, τη μεταφορά 149 Ασσυρίων στη Σλοβακία. Οι Ασσύριοι είναι οι τελευταίοι που μιλούν τα αραμαϊκά, τη γλώσσα που μιλούσε ο Χριστός. Υποστηρίζω το ψήφισμα. Ευχαριστώ κύριε Μαμίκινς. Από ό,τι φαίνεται η κυρία Σαπόρσκα είχε ζητήσει, ε, χάθηκε η αίτησή για την επεξήγηση. τη δίνω όμως το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Διεθνές Δίκαιο έχει θεσπίσει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια σήμερα με τα οποία χαρακτηρίζεται μια πράξη σαν γενοκτονία και πρόκειται επομένω για κάποιε πράξει οι οποίε έχουν ως σκοπό να εξοντώσουν μια εθνότητα ή ε, κάποιους που έχουν την, ίδια θρησκεία και οπότε πράξεις αυτές αποσκοπούν στην ε, καταστροφή, στην εξόντωση κάποιων και αυτό γίνεται στην ε, Συρία και στο Ιράκ με τους χριστιανούς άρα τον πούμε ότι αυτό είναι γενοκτονία αυτό είναι το πρώτο βήμα ούτως ώστε το θέμα να πάει στο Συμβουλίο Ασφαλείας και να επιληφθεί το Διεθνές Δικαστήριο επομένως θα πρέπει ε, επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ε, κάποια συγκεκριμένη θέση, κάποιον αξιωματούχο ο οποίος να ασχοληθεί με τα δικαιώματα των χριστιανών και των άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων σε όλο τον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι εγκρίθηκε αυτό το ψήφισμα το οποίο θα είναι κείμενο ιστορικό για το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαπόρσκα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτό το θέμα, τελειώσαν η επεξηγής ψήφου. Καλή σας όρεξη. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3. Καλή όρεξη σε όσους είναι ακόμα παρόντες.